afterwards. everyone. Καλώς, καλησπέρα σε όλους. Συνήθεια το έχουμε κάνει να συνεδριάζουμε στο Στρασβούργο. Δεν θα σας ρωτήσω πώς το βλέπετε, εν πάση περιπτώσει. Χαίρομαι εγώ που σας βλέπω. Ε, αν είστε εντάξει με την ημερήσια διάταξη, να θεωρούμε ότι εγκρίθηκε στις 6 Δεκεμβρίου, που είναι και του Αγίου Νικολάου, ημέρα Πέμπτη, Είχαμε προβλέψει ε, να την κρατήσουμε αυτή την ημερομηνία, μήπω έχουμε συνεδρίαση το απόγευμα, αλλά τώρα μπορώ να σας πω ότι δεν θα συνεδριάσουμε. Στις 20 Νοεμβρίου έχουμε ανταλλαγή απόψεων με το Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το δικαίωμα στην υγεία. στα πλαίσια της Εβδομάδας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που διοργανώνεται για να γιορτάσουμε την 70η επέτειο της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα έχουμε ανταλλαγή ε, απόψε με τον δόκτωρα Τέντρο Σαντάνομ Γκεμπρεγέσους που είναι Γενικός Διευθυντής του ΠΟΕ, ΠΟΗ. Έχουμε και τον Κούτελαν τον ε, νεότερο απόψε εδώ μαζί μας. 5 ε, με 6 το απόγευμα. Ε, παρακαλώ, ελάτε. Είναι ο γιος Ελάτε σας παρακαλώ. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, είναι ανοιχτή στη συνεργασία με σημαντικούς θεσμούς και οργανισμούς όπως είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Και το δικαίωμα στην υγεία είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες. Μας παρακαλώ λοιπόν να έρθετε γιατί θα σας ενδιαφέρει και εσάς. Είναι πολύ μικρή σε διάρκεια ανταλλαγή απόψεων, μία, μία ώρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και μετά μια σύντομη δεξίωση, 6 και μετά. Έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες για τη συνεδρίαση αυτή και ως συνήθως μεταδίδεται στο διαδίκτυο και έχετε λάβει και το φάκελό σας από το διαδίκτυο. We did that. Okay, so that's, uh, then uh, we can move. Ωραία, μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Πάμε αμέσω. Πρώτη ψηφοφορία είναι για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ. Αρχίζουμε. Τροπολογία 88. Ψήφι υπέρ. Α, όχι, δεν την ψηφίζουμε. Γράφει εδώ. Ζητώ συγγνώμη. Ωραία, αρχίσαμε. Ζητώ συγγνώμη. 89. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 92 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Με 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Όχι. 111. Εγκρίθηκε. 109. αλλά δεν ψηφίζουμε την 110 γιατί καταπέπτει. Παρ' όλα αυτά, κύριε Γκίζε, και από ό,τι είδα, σας υποστηρίζουν στην πρότασή σας. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 131 και 132 υπέρ κατά καταπίπτων 129 was rejected. Okay. 129 απερίφθη. 131-132 ε, μαζί. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 135 Θέλετε έλεγχο την 134 να επαληθεύσουμε. Ας την επαληθεύσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Από το ΕΛΚ για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. <laughs> Ευχαριστώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μικρή διαφορά. Οι φιλελεύθεροι φταίνε που δεν λένε τι ψηφίζουν. 135 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. Αρχίζει τώρα η υπολήθευση. Πέρας. Απόρριπτεται. 141 υπέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 142 υπέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 143 υπέ. Κατά. Αποχές έλεγχος παρακαλώ. 143 αρχίζει τώρα. Πέρασε. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το έλκτη υπέρ ή κατά. Ε, εγκρίνεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Για είναι 148 ελέγχου αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. And is closed. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. Ε, 149 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 17 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 176 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, έλεγχο παρακαλώ. 176 πολυθεύουμε, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. και τελειώνει. Και εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά έλεγχος. 180 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 182 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 183 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 184 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 186 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 185, όχι συγγνώμη, 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 188 in favor. 188 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 189 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 190 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 191 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 192 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 193 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος. 194 αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Εγκρίθηκε. 195 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 207 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 209 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία στην 25 τροπολογία. Νομίζω ότι είχε εγκριθεί, αλλά για καλό και για κακό, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίθηκε. 26 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 28 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Αν θέλετε μπορούμε να την ελέγξουμε, θέλετε. 28 αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Δεν σηκώνετε χέρια, αλλά ε, περίμενα τον κύριο Γκερμπράντι να μας πει τι κάνουν φιλελεύθεροι πέρας. απορρίπτεται. Οι φιλελεύθεροι δεν σηκώνουν χέρια. Λοιπόν, 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η 40 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 47 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 52 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος. Παρακαλώ τσακάρουμε την 53, αρχίζει τώρα η ηλεκτρονική απολύθευση. Πέρασε. Απορρίπτεται. 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 και 56 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 72 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 76 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 77 όχι, 78 υπέρ, κατά αποχές Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 78, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. And it's Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 81 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 82 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 83 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 84 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 85 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα. Ωραία. Πέρες. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η επόμενη ψηφοφορία. Which 120? την πρόταση κανονισμού θέσμιση του προγράμματος συμβεστιού. Του κυρίου Μπέλετ. Έτσι ακούγεται. Έτοιμος, έτοιμη εντάξει. Αν φτάνουμε στις συμβασμούς 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές καταψήφισαν οι σοσιαλιστές. Ας ελέγξουμε γιατί δεν είμαι απολύτως σίγουρη. 67 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 84. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και πέρας. Και εγκρίνεται. Για μία ψήφο. Κυρία Ικχάουτ. Ωραία, ωραία. Ευτυχώς που είσαστε παρόν και υπερψηφίσατε τη δική σας τροπολογία. Λοιπόν, 97 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α, ας ελέγξουμε. 99 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά ελέγχουμε την 105 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Λόγω ισοψηφίας. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 109 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 110 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 111 υπέρ, κατά αποχές ελέγχουμε την 111. 111 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 προφορική. Υπάρχει κάποιος που αντιτάσσεται στην προφορική που έχετε στον κατάλογο. Εάν όχι, ψηφίζουμε μαζί με την προφορική υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά αποχές. Τι κάνει Γκουε, πώς ψηφίζει, υπέρ. Τότε ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν ψηφίζετε όλοι, αλλά δική σας επιλογή. Είμαστε 49 παρόντες και μόνο 46 έχουν ψηφίσει. Ωραία, πέρασε. Ισοψηφία, βλέπετε. Άρα αυτοί που δεν ψήφισαν θα έκαναν τη διαφορά, άρα απορρίπτεται. Λοιπόν, 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 122, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές Ελέγχουμε την 127. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Τι κάνει κουέ. Δεν βλέπω καμία ένδειξη. Άρα ελέγχουμε την 128. Άρχεται. Πέρας. Και απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 129. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά υπέρ της 132 υπέρ κατά ελέγχουμε την 132 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Και εγκρίνεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δύσκολα, δύσκολα απόψε. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά Ας ελέγξουμε καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Έχει κανείς λίγη σοκολατίτσα, κάτι. Όχι, όχι η ζάχαρη. Ε, εγκρίνεται λοιπόν. 142 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 152 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται.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 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 57 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά, άρχεται. And it is uh, nearly closed. Πέρας, σχεδόν πέρας, πέρας και εγκρίνεται. Bravo. Okay. Μάλιστα. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία της γνωμοδότησης για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027. Τροπολογία 24. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφέ το αποτέλεσμα. Στο ψηφίσουμε, στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία για την 25. And it's closed. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 26. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Αν ψηφίζετε έτσι που να καταλάβω. Είναι περίεργο. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία.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 κατά. Οι σοσιαλιστές τι είναι, υπέρ ή κατά. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για τη 45. Καλώς. Άρχεται ηλεκτρονικά η ψηφοφορία για τη 45. Τέλος. Απορρίφθηκε. 46. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 47. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται που είμαι α, 48 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επτά υπέρ κατά αποχές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 κατά αποχές εγκρίνεται. Την 23 δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και φτάσαμε στο τελευταίο θέμα της ψηφοφορίας. Τελευταίο δεν είναι. Μάλιστα. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του διαστημικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινάμε με τροπολογία 59. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 61. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64 και 52 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνονται. 65. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 66. Υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 67. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 και 76 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αν επιμένετε, αλλά πείτε μου μέχρι πού. 78 με 83 πρώτα να ψηφίσουμε μαζί. Α, δεν μπορούμε γιατί είναι διαφορετικέ ενδείξει. Θα τα περάσω γρήγορα πάντω. 77, 77. Θα είμαι γρήγορη. 77 Ποιο είναι υπέρ κατά αποχέ. απορρίπτεται. 78 υπέρ κατά αποχέ. απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται, 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 84 υπέρ α, κατά αποχές εγκρίνεται. 85 ποιος είναι υπέρ Ποιο θέλει ηλεκτρονικό έλεγχο για την 84, το ΕΛΚ. Πολύ ευχαρίστω. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 84, ηλεκτρονικό έλεγχο. Τέλο ψηφοφορία. Έγκρινεται. 85, ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά αποχέ. Απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά αποχέ. Απορρίπτεται. 88 και 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 89 και 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 90 και 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και θα έχουμε ένα σύνολο τροπολογιών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 και 46 υπέρ κατά αποχές εγκρι... απορρίπτονται 105 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Μπορούμε πάλι να ψηφίσουμε μαζί κάποιες τροπολογίες. Η πράσινη λέει πρώτα μέχρι το 121 τότε, αν θέλετε μαζί ψηφοφορίες. Από την, 100, ε, από την 106 μέχρι την 121, συμφωνείτε, να ψηφίσουμε μπλοκ. Όχι, το ECR διαφωνεί. 106 με 111. 106 με 111 ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 112 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ. Μπορούμε να ψηφίσουμε τις 113 με 121 μαζί. Αν συμφωνούμε όλοι. Και το ECR συμφωνεί, οπότε ψηφίζουμε τις τροπολογίες 113-121. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μπορούμε και πάλι να ψηφίσουμε μαζί μερικές τροπολογίες Καλώς ξεχωριστά. 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τώρα 126, γιατί υπάρχει διαφωνία εδώ απόψε. Ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Εντάξει, εντάξει. Κύριε δεν ελπίζω να ξέρετε τι κάνετε. Γιατί σας κοιτάζα όταν είπα ότι απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται ψηφοφορία για την 126, τέλος. Α, εγκρίνεται. Πότε μπορώ να στηρίζομαι σας. Εγκρίνεται λοιπόν. 132 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 132, γιατί εγώ θα έλεγα ότι απορρίπτεται, αλλά δεν μπορώ να είμαι και βέβαια Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Όντως απορρίπτεται. 133. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται.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 κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 150 άρχιτη ψηφοφορία And is closed. τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά αποχέ απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά αποχέ απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά αποχέ απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά απόχέ, απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά αποχέ απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά αποχέ απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά απόχέ. εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 27 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 31 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 32 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 33 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 34 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 36 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 37 υπέρ, κατά αποχές,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 Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχο για την 54. Άρχεται η ψηφοφορία. What is on 54? Thank you. And it is a Τέλος. Εγκρίνεται 54. Εγώ τι είχα πει. λυπάμαι. 55. ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά παρακαλώ άρχεται ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίθηκε ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες σας ευχαριστώ πολύ και κυρίως και το πέρα συνεδρίασης καλό βράδυ καλή όρεξη Ραντεβού αύριο. Γεια σας.